εγκρίνεται. Μέρος δεύτερο υπέρ, κατά, αποχές, να το επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Συγγνώμη. Ψηφίζουμε το δεύτερο μέρος της 15. Μέρος δεύτερο. Και πέρας και έχει απορριφθεί. 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία και πέρασε. και εγκρίνεται σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας εγγυώμαι ότι πολλοί πολίτες θα ικανοποιηθούν για αυτήν την ισχυρή έντολη σας ευχαριστώ. Τελειώσαμε με τις ψηφοφορίες. Όσοι σκοπεύετε να φύγετε, παρακαλώ ησυχώ για να περάσουμε στο επόμενο θέμα σε λίγα λεπτά. So, now when people... Λοιπόν, τώρα που έφυγαν όσοι ήθελαν να φύγουν, περνάμε στο σημείο 15, αναφορά 63 08 και 0408 όσον αφορά η καζόμενη παραβίαση δικαιωμάτων των καταναλωτών στις διαδικασίες διαταγής πληρωμής στην Βουλγαρία. Είναι εδώ, είναι στο κτίριο. Αναφέρονται αλλά δεν ε, έχουν έρθει ακόμα. Σε 15 λεπτά. Ε, δεν μπορείτε να, να, να τους περάσετε μπροστά από την ουρά. Now there is someone coming. But there are three different ones and um, okay, but we, we Is there someone coming now? Έρχεται κάποιος τώρα για μία από τις αναφορές. Okay. The next item. Let's see if we can deal with that. Do I have from... Λοιπόν, υπάρχει ο κύριος Γαβριλιάδης από την Κομισιόν. Ωραία. Πάμε λοιπόν στο σημείο 16. η 10-15 για το θέμα της ελευθερίας έκφρασης και της καταστολής ε, των δημοσιογράφων στη Μάλτα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αλλά ο συνάδελφός μου δεν έχει έρθει γιατί υπάρχει και το θέμα της ελευθερίας ε, έκφρασης και μιμιέ. βεβαίως μπορώ να καλύψω ε, μέρος, αλλά όχι και τα δύο μέρη. Να, σα καλύψουμε το δικό σας και να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, να ξεκινήσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και σβήνει το μικρόφωνο του Μιλτή. αναφορά φύγει κάποια ζητήματα που αφορούν την τρέχουσα κατάσταση στην ε, Μάλτα. Ε, βεβαίως όλα ξεκίνησαν από την ε, δολοφονία, την φρικτή στην Μάλτα. Η Κομισιόν είχε διάφορες ευκαιρίες, είχε εκφράσει την ανησυχία της για την κατάσταση. Καλέσαμε την κυβέρνηση Μάλτας να κάνει ό,τι μπορεί να διερευνήσει το έγκλημα, να οδηγηθούν οι δάστες στην δικαιοσύνη. Η Επιτροπός Γιούροβα είχε πάει εκεί την προηγούμενη εβδομάδα και επανέλαβε ακριβώ αυτά τα πράγματα στην κυβέρνηση της Μάλτας και στην Υπουργό Δικαιοσύνης όσον αφορά τα γενικότερα ζητήματα για το κράτος δικαίου. Η Κομισιόν είχε την ευκαιρία να το θίξει προφορικά αλλά και στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου το οποίο όπως όλοι γνωρίζουμε είναι ακριβώς το εξάμεινο συντονισμού της οικονομικής πολιτικής των κρατών μελών Φέτος λοιπόν υπάρχει ένα συγκεκριμένο κομμάτι στην έκθεση για την Μάλτα που δημοσιεύτηκε τον Μάρτιο που αφορά ακριβώς ε, την δικαιοσύνη και την αναποτελεσματικότητα του συστήματος που αναφέρεται στην διαφθορά ε, να σας πω ότι η διαφθορά είναι ευθύνη του Επιτρόπου Αβραμόπουλου και βεβαίως ε, ζητήματα ξεπλήματος χρήματος και μετά η Κομισιόν ενέκρινε και συστάσεις συγκεκριμένες με συγκεκριμένη αναφορά σε ζητήματα ξεπλήματος χρήματος στην Μάλτα και με αναφορά στο αναποτελεσματικότητα του συστήματος ε, της δικαιοσύνης. Ε, η Επιτροπός Γιούροβα ήρθε από τη Μάλτα πριν από τρεις μέρες. Αυτά για την ώρα όσον αφορά την ελευθερία έκφρασης θα προτιμούσα να σημερώσουν οι συνάδελφοι βεβαίω από τη Γενική Διεύθυνση Connect. Σας ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ που είστε τόσο ευέλικτος. Έχει έρθει ο συναδελφός σας, όχι. Η κυρία Μπαλσέλς από την Connect, όχι. σας δώσουμε λοιπόν τον λόγο στους βουλευτές. Θέλει κάποιος τον λόγο. Ναι. Ακριβώς. Μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι το κοινοβούλιο έχει ήδη κάνει πολλά πράγματα. 15 ε, Νοεμβρίου ε, περάσαμε ένα ψήφισμα και στείλαμε μια διπροσωπη ad hoc στη Μάλτα το τέλος του περασμένου έτους ε, και αυτό το οποίο συμβαίνει, είτε μιλάμε για τη Μάλτα είτε για οποιαδήποτε άλλη χώρα. Αυτό το οποίο συμβαίνει βεβαίω ενδιαφέρει ολόκληρη την Ένωση. Το κράτος δικαίου είναι αντικείμενο συλλογική ε, εξέταση. Η δολοφονία της κυρίας ε, Γκαλίτσια ακριβώ στόχο είχε να ε, ενσπείρει τον φόβο όπως αναφέρει το ψήφισμα, ε, ειδικά σε όσους ερευνούν περιπτώσεις διαφθοράς ε, και εξεπλήματο χρήματο. Έγιναν λοιπόν διάφορες ε, παραστάσει στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Νομίζω λοιπόν ότι όλοι μπορούμε να εκφράσουμε την λύπη μας για τα όσα συνέβησαν στην ίδια, στην οικογένειά της για να εκφράσουμε τα συλληπιτήριά μας. Κάποιος άλλος θέλει να πει κάτι. Πίτερ. Θα ήθελα να πω κάποια πράγματα γιατί α, τα είπε η πρόεδρος τα συνόψισε καλά πρέπει να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά όταν ε, πρέπει να διερευνηθούν τέτοια πράγματα αν γίνουν ε, σωστά αυτά τα πράγματα νομίζω ότι υπάρχει και μία φάση ε, σιωπής. Εμείς ε, παρόλα αυτά και μια φάση ησυχία. Ε, εμείς ε, παρόλα αυτά θεωρούμε ότι πρέπει να παραμείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά ως έκφραση θλίψης αλλά και πολιτικής βούλησης ότι πρέπει δηλαδή να διερευνηθούν 100% τα συμβάντα αυτά. Εντάξει, να γίνει σωστά η δουλειά και όχι γρήγορα, αλλά να μην δημιουργείται η εντύπωση ότι υπάρχει εδώ πέρα κάποια καθυστέρηση. Πριν από αυτό το περιστατικό ε, θα ορκιζόμουν ότι δεν μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πραγματικά ήταν αδιανόητο. Γιατί πραγματικά ε, θεωρώ ότι θα έπρεπε να έχει σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για σε άλλε εποχές. Σας ευχαριστώ Πίτερ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι μπορώ να το συνοψίσω ε, και χωρίς ε, τον συνάδελφό σα κύριε Καβριλιάδη. Κύριε Κοσολίνη, θέλετε να μιλήσετε. Ναι, ακριβώς για τους λόγους που μόλις άκουσα. Εγώ θα πρότεινα αντιθέτω να κλείσει αυτή η αναφορά και θα αποστείλω στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ και στον ε, αρμόδιο επίτροπο το αίτημα να μας ε, ε, κρατούν ενήμερους και ακριβώς λόγω της φύσης των αιτημάτων. Και μάλιστα πρόκειται ο ετών είναι κάποιος Βερτανός που ζει στις Ηνωμένε Πολιτείες και κάνει μια αναφορά ε, σαν να μην ξέρει ακριβώς ε, το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην ε, Μάλτα για τα γεγονότα τα οποία αφορούν την τρομερή αυτή υπόθεση. Θα σας πρότεινα λοιπόν κάτι το συγκεκριμένο και μία αναφορά λιγότερο γενικόλογη. αλλά το να την κλείσουμε επειδή είναι και πολύ γενικόλογοι μου φαίνεται και κάπως ε, ε, μια εργαλειακή χρήση και για πολιτικούς σκοπούς. Λοιπόν, η ίδια επίτροπος η οποία είχε πάει στη Μάλτα τις ε, προηγούμενες εβδομάδες και Νομίζω ότι ακριβώς θα πρέπει να περιμένουμε λίγο τα αποτελέσματα, αλλά το να κλείσουμε την αναφορά δεν ξέρω, μου ακούγεται κάπως ε, πολιτικό ζήτημα και θα πρέπει να πούμε λίγο και στην ουσία. Ευχαριστώ, Σεσίλια. που αναφέρθηκε η Λίμπε, να πω τώρα ότι η γεγονός είναι ότι η Λίμπε έχει αναλάβει το θέμα. Όπως ξέρετε υπάρχει μια ομάδα κράτους δικαίου που παρακολουθεί την κατάσταση σε Μάλτα και Σλοβακία και ακριβώς θα εξετάσουμε όλα αυτά τα στοιχεία που μόλις αναφέρθηκαν από τους εκπροσώπους της Κομισιόν αλλά για αυτόν ακριβώς το λόγο θέλω η αναφορά αυτή να παραμείνει ανοιχτή στην Επιτροπή αυτή γιατί αν δείτε τις διάφορες επιτροπές που έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για να σχοληθούν μετά τις ΛΥΒΕ θα έλεγα ότι η Επιτροπή μας που εκπροσωπεί όλους τους πολίτες και εδώ μπορούν να προσέλθουν όλοι οι πολίτες από οποιοδήποτε κράτη-μέλος ανεξαρτήτως του που ζουν Βλέπουμε εδώ πέρα λοιπόν πάρα πολλές λεπτομέρειες από τον συγκεκριμένο αναφέροντα, είναι πολύ ακριβής. Θα έλεγα λοιπόν ότι η Επιτροπή Αναφορών, ειδικά η Επιτροπή μας, είναι αυτή η οποία θα πρέπει να ε, ανησυχεί και να εμπλακεί αυτό το ζήτημα γιατί οι Μαλτέζοι όπως ακούσαμε από τους συναδέλφους μας κοιτούν πολύ προσεκτικά το τι συμβαίνει. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θέλω και εγώ να αντιδράσω στην ε, τοποθέτηση του συναδέλφου. Είμαι υπεύθυνο από πλευρά του ΕΛΚ ε, όταν ήμουν στη Λίμπε, στηρίζω όλες τις δραστηριότητε της Λίμπε. Είναι πάρα πολύ καλό. Εγώ είμαι Σλοβάκος ε, πολίτης, οπότε φυσικά και με απασχολεί το θέμα και θέλω να είμαστε δραστήριοι. Το ΕΛΚΟ όμω είναι σαφώς κατά της ε, στήριξη του να μείνει ανοιχτή. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να παρακολουθήσει τις δραστηριότητες όχι μόνο των μαλτέζικων αρχών αλλά και των ευρωπαϊκών. Η κυρία Μίση. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Πριν συνεχίσουμε τη συζήτηση αυτή που είναι βέβαια πάρα πολύ σημαντική, θα θέλω να αναφέρω κάποια γεγονότα. Πράγματι, πρέπει να είμαστε αντικειμενικοί. Και να μην ξεχνάμε ότι η αναφορά αυτή υποβλήθηκε λίγες μόνο μέρες μετά το φοβερό έγκλημα κατά της, της κυρίας Γαλίτσια και πολλά πράγματα έγιναν έκτοτε. Πρέπει να καταλάβουμε ότι οι αρχές της Μάλτας έχουν ε, κάνει κάθε προσπάθεια έτσι ώστε να υπάρξει πλήρης διερεύνηση και να μην μείνει τίποτα χωρίς να ερευνηθεί. FBI, Interpol, όλοι κλήθηκαν μετά το έγκλημα αυτό. Οπότε μέσα σε τρεις εβδομάδες οι ύποπτοι για το έγκλημα αυτό ε, συνελήφθησαν και διερευνείται η υπόθεση. Αυτό είναι γεγονός. Δεν μπορούμε να περιμένουμε βέβαια να παραμένει το ζήτημα για πολύ. Πρέπει όντως να καταλήξουμε στη δικαιοσύνη γρήγορα για το θύμα, για την οικογένειά του, αλλά και για όλους μας. Οι δράσεις τώρα που ανέλαβε η κυβέρνηση δεν είναι δράσεις κυβέρνησης η οποία παραβλέπει το κράτος δικαίου, αλλά μια κυβέρνησης η οποία θέλει να φτάσει μέχρι το τέλος την έρευνα αυτή για το έγκλημα που σόκαρε ολόκληρη την Ευρώπη. Θέλουμε και εμείς υπεύθυνοι να πάνε στη δικαιοσύνη όσο γίνεται πιο γρήγορα. Άρα δεν πρέπει να κατακρίνουμε το κράτος δικαίου στη Μάλτα. Τώρα, σε σχέση ακριβώ με το κράτο δικαίου, συζητήθηκε δύο φορέ στην Ολομέλεια και με το Σεβούλιο και με την Επιτροπή που εκφράστηκαν δημόσια και πολλέ άλλε φορέ σε διάφορε επιτροπέ. Διερευνητικέ ε, αποστολές, αντιπροσωπείες πήγαν για να δουν τι γίνεται με το κράτος ε, δικαίου στην ε, Μάλτα τι έγινε με τη διερεύνηση του εγκλήματος αυτού κατά της κυρίας Καλήθεια. Από εκεί και πέρα το κράτος δικαίου υπάρχει σε όλες τις χώρες μέλη και είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην γίνεται καμία παραβίαση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξετάζει την τρέχουσα κατάσταση στη Μάλτα έτσι αλλιώς. Και πρέπει να σας πω ότι δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα με αυτό του να εκτιμά και να αξιολογεί την αναφορά αυτή. Ο να έχει κάθε δικαίωμα να την υποβάλει. Το ερώτημα όμω είναι αυτό πρέπει να γίνεται από κάθε κοινοβουλευτική επιτροπή. Μην το ξεχνάμε, όπως έχει διποθεί, ότι η ΛΥΜΠΕ είναι η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή. Και η ΛΥΜΠΕ ήδη δουλεύει πάνω σε όλα τα ζητήματα τα οποία θίγει και αναφέρον στην αναφορά του. Οπότε γιατί δεν υπάρχει επικάλυψη. Υπάρχουν τόσες πολλές αναφορές που μας περιμένουν να τις εξετάσουμε και είναι αρμοδιότητα της δικιάς μας Επιτροπής. Επιπλέον, ο Υπουργός Δικαιοσύνη τη Μάλτας δέχτηκε την πρόσκληση της Λίμπε να έρθει και να απαντήσει στι ερωτήσει τη. Αρμόδια επί τη ουσία είναι η ΛΥΜΠΕ, λοιπόν, και αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μα. Τέλο, αλλά όχι και λιγότερο σημαντικό, Πρόσφατα η Υπηρεσία Οικονομικών Πληροφοριών εμφάνισε, είπε ότι πρόκειται για μία από τις 11 χώρες που έχουν πλήρη δημοκρατία και ότι που ζητάει επίσης την αξιολόγηση των παραβιάσεων. Πέρα από όλα τα γεγονότα τα οποία ανέφερα μέχρι τώρα, που είναι γεγονότα, έτσι, δεν είναι προπαγάνδα, η σύστασή μου είναι να κλείσει η αναφορά αυτή. Περισσότερα από τα θέματα που θίγει ο αναφέρον έχουν ήδη αντιμετωπιστεί για τα άλλα, τα έχει αναλάβει είτε η Λίμπε, είτε οι αρχές της Μάλτας. Γι' αυτό λοιπόν και ζητάω η αναφορά αυτή να κλείσει, κυρία Πρόεδρε. Πρόεδρο, σε ευχαριστούμε. Η κυρία Ντάλη έχει ζητήσει το λόγο επίσης. Παρακαλώ. Πολύ σύντομα. Πρώτα απ' όλα, να κάνουμε τη δήλωση ότι επιβεβαιώνονται υποθέσεις είναι σαν να καταλήγουμε πολύ γρήγορα σε συμπεράσματα δεδομένου ότι συνεχίζονται οι έρευνες και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξετάζει το ζήτημα σε βάθος. Και δεν πρόκειται μόνο για ένα θέμα της Μάλτας, γιατί όπως ακούσαμε ήδη, μάθαμε ότι υπάρχει και άλλη δολοφονία στη Σλοβακία, άλλου δημοσιογράφου. Οπότε το ζήτημα πηγαίνει πολύ περισσότερο σε βάθος. Όμως θα ήθελα να ζητήσω από την Επιτροπή μας να κλείσει αυτή την αναφορά. Γιατί εμείς δεν λέμε ότι θέλουμε να κλείσει το ζήτημα. Φυσικά και δεν θέλουμε να κλείσει. Ήμασταν ξεκάθαροι σε αυτό και στην αρχική μας αντίδραση απέναντι στον αναφέροντα. Όμως όλοι γνωρίζουμε ότι συνεχίζεται δουλειά, συνεχίζονται οι έρευνες, η ΛΥΜΠΕ δουλεύει πάνω σε αυτό το θέμα και στη Μάλτα οι αρχές βάσει του κράτους δικαίου και στη Σλοβακία επίσης. Και σίγουρα θα υπάρξει και άλλη αντιπροσωπεία που θα κοιτάξει τις λεπτομέρειες. Συνεπώς, θέλω να σας ζητήσω να ακούσετε την πρόταση που έγινε, δηλαδή η Επιτροπή μας να κλείσει αυτή την αναφορά. Πάντα όμως μπορούμε να ζητήσουμε από την ομάδα εργασίας να μας ενημερώνει για τις εξελίξεις δεδομένου μάλιστα που θα συνεχιστεί αυτή η δουλειά. Αν αφήσουμε ανοιχτή αυτή την αναφορά, υπάρχει επικάλυψη στο έργο μας εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρόεδρος, εύκολα μπορεί κανείς να συνοψίσει νομίζω. Τέλος πάντων, θα προσπαθήσω. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται όντως η Επιτροπή κάτι να προσθέσει. Είναι πολύ πολιτικό το θέμα, έτσι πρότασή μου θα ήταν να κρατήσουμε ανοιχτή την αναφορά, να τη στείλουμε στη ΛΥΜΠΕ, στην ομάδα εργασίας που ελέγχει τα περί κράτους δικαίου, να εξηγήσει ο αναφέρον κτλ. Και, να ζητήσουμε από τη ΛΥΜΠΕ επίση, αν έχει ακροάσεις ή άλλες σχετικές δραστηριότητες, να μας συμπεριλάβει, ώστε να μπορούμε και εμείς να επωφεληθούμε και να συνεισφέρουμε και εμείς που έχουμε τις αναφορές των πολιτών και να σταλεί και επιστολή στη Βεραγιούροβα η οποία επέστρεψε από αποστολή που πήγε πρόσφατα και να παραμείνει ανοιχτή αναφορά. Γιατί σίγουρα θα προχωρήσει το σώμα για αυτό το ζήτημα. Υπάρχει όμως άλλη πρόταση που λέει να κλείσει η αναφορά αυτή. Οπότε, ποιος θέλει να ακολουθήσει τη δικιά μου σύσταση για το πώς θα συνεχίσουμε. Πρέπει να το μας το δείξετε καλά, έτσι, σηκώστε χέρια. Επτά. Και ποιοι είναι υπέρ της πρότασης της κυρίας Μίτση, να κλείσει δηλαδή αναφορά. Τέσσερις. Πέντε. Ωραία, ψηφίσαμε. Έχουμε απόφαση. Παραμένει ανοιχτή λοιπόν. Και θα κάνουμε αυτά τα οποία σας ανέφερα. Και τώρα νομίζω ότι μπορούμε να αφήσουμε αυτό το θέμα σήμερα και να επιστρέψουμε στο σημείο 15 που είναι τρεις αναφορές για εικαζόμενη παραβίαση των δικαιωμάτων των καταναλωτών στις διαδικασίες διαταγής πληρωμής στη Βουλγαρία και πρόκειται επίση και για ένα πρόβλημα όσον αφορά τα ανυπόθηκα δάνεια. Έχουμε τρεις αναφέροντε εδώ μαζί μας. Σας καλωσορίζουμε όλους. Καλώς ήρθατε. Θα σας δώσουμε το λόγο. Τρία-τέσσερα λεπτό καθένας. Έτσι, γιατί πρόκειται για το ίδιο ζήτημα βασικά. Οπότε ο κύριος Ήλιεφ, παρακαλώ μετά η κυρία Ντεσλάβα Φιλίποβα και τέλος η κυρία Βιολέτα Γασποντίνοβα. Βέβαια εσείς μπορείτε να αποφασίσετε με ποια σειρά θα πάρετε το λόγο για να μας παρουσιάσετε τα θέματά σας. Τρία-τέσσερα λεπτά ο καθένας παρακαλώ, έτσι. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρίες και κύριοι. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο απασχολεί πολλούς ε, Βούλγαρους ε, πολίτες και τους έχει καταστρέψει οικονομικά. Οι τράπεζες στην χώρα έχουν προνόμιο, δηλαδή πρακτικά μπορούν να να προχωρήσουν ε, σε μια εκτέλεση μέσω των δικαστηρίων και δεν υπάρχει δυνατότητα προσφυγής ε, από τους ε, αντιδίκους. Ουσιαστικά τα δικαστήρια έχουν γίνει ε, απλοί εκτελεστές ε, της θέλησης ε, των τραπεζών. Υπάρχουν καταχρηστικές ρήτρε στις δανειακές συμβάσεις και επιπλέον τα δάνεια αυτά επίσης υπολογίζονται σε ελβετικό φράγκο και συχνά οι καταναλωτές ε, μετά από μακρόχρονη διαδικασία λαμβάνουν πίσω την περιουσία τους αλλά εντωμεταξύ έχει αυτή εκπληστηριαστεί ε, το, το πραγματικό ακίνητο δηλαδή και πολλοί πολίτες γι' αυτόν τον λόγο αναγκάζονται να μεταναστεύσουν και στο εξωτερικό. Καλημέρα και από μένα. Ναι δικηγόρος. Έχω ασχοληθεί με αυτά τα ζητήματα γιατί με έχουν πλήξει και προσωπικά. Το σημαντικότερο θέμα εδώ είναι ότι το κράτος ουσιαστικά έχει εκχωρήσει την κυριαρχία του στις τράπεζες. Δηλαδή τα δικαστήρια απλά καταγράφουν την θέληση των τραπεζών ε, και οι τράπεζες έχουν γίνει, έχουν καταστεί σαν ένας καρκίνος στο σώμα της κοινωνίας, ένας καρκίνος που έχει κάνει μετάσταση σε διάφορες ε, πόλεις. Μόνο δικαιώματα έχουν, υποχρεώσεις δεν έχουν και έχοντας αυτά τα προνόμια να κάνουν ό,τι θέλουν δηλαδή, ε, τελείως αυθαίρετα πραγματικά κάνουν ό,τι θέλουν. Ε, οι αναγκαστικέ εκτελέσει στη Βουλγαρία λαμβάνουν χώρα χωρί άλλε συνθήκε. Χωρί να ενημερώνεται ο φιλέτη καν. Γιατί υπάρχει ε, αυτή η δυνατότητα, αυτά τα απίστευτα προνόμια που δίνει ο νόμος της ε, τράπεζας. Δεν χρειάζεται καν να ενημερώσουν τον ενδιαφερόμενο. κάποιος να μηνυθεί χωρίς να ενημερωθεί καν. Ε, έχουμε λοιπόν θέσει το ζήτημα αυτό και στη Βουλγαρική Βουλή εδώ και χρόνια. Οι τράπεζες έχουν μια μονοπωλιακή θέση. Καθορίζουν τα επιτόκια όπως θέλουν και το δικαστήριο δεν έχει δικαίωμα να τοποθετηθεί επί του θέματος. Ο νόμος ε, δίνει δικαιώματα μόνο στις ε, τράπεζες. Οι καταναλωτές ε, δεν γνωρίζουν ότι μπορεί να κάνουν κάτι όταν αλλάζουν τα επιτόκια, επιβάλλονται τιμωρητικοί τόκοι χωρίς όρια. Είτε μέσω των εταιριών τους, είτε μέσω ενδιαμέσων, αγοράζουν την ε, περιουσία των οφειλετών οι τράπεζες ε, και εκμεταλλεύονται την θέση των οφειλετών και μια τελευταία παρατήρηση οι τράπεζες δεν αναλαμβάνουν κανέναν κίνδυνο ε, μπορείτε να συντομεύετε παρακαλώ ναι σας ευχαριστώ θα σας τα δώσω και έγραπτος Ωραία. Και τώρα ο κύριος Ήλιεφ. Καλημέρα σας ε, κυρίες και κύριοι ευρωβουλευτές. Είμαι εκπρόσωπος μιας πρωτοβουλίας ε, πολιτών μιας ένωσης ε, στη Βουλγαρία που στόχο έχει να προστατεύσει τα δικαιώματα των καταναλωτών, των οφηλετών στην Βουλγαρία. Το θέμα δεν είναι μόνο εθνικό. Είναι υπερεθνικό θα έλεγα. Το θέμα αφορά και Ολλανδούς και Γερμανούς καταναλωτές ε, που εντωμεταξύ έχουν ε, δικαστεί και καταδικαστεί έχουν υπάρξει πληστηριασμοί της ιδιοκτησίας τους. Σχεδόν η μισή Βούλγαροι πολίτες, μιλάμε για εκατομμύρια ανθρώπους, ε, πλήττονται πλέον από αυτήν την υπόθεση. Το δικαστήριο δεν κάνει κάποιον έλεγχο εξοφίτσιο για τα αιτήματα πληρωμής των ε, τραπεζών. Ε, έτσι δηλαδή δεν ε, συμμορφώνεται με την οδηγία 93 κάθετος 19 που αφορά τις καταχρηστικές ρήτρες πάνω από 300.000 ε, τέτοιες ε, περιπτώσεις έχουν υπάρξει τα τελευταία χρόνια και δεν ε, έχουν ακόμα καταλήξει κάπου. Εν τω μεταξύ τα... η περιουσία έχει εκπληστηριαστεί και οι τράπεζες τελικά είναι μια εγκληματική οργάνωση που ακολουθεί διεφθαρμένες πρακτικές ε, σε συνεργασία με τα δικαστήρια τα βουλγαρικά. Υπάρχουν ε, επίσης ε, γύρω στους 600 δικαστικούς κλητήρες και 200 ιδιώτες επίσης οι οποίοι είναι αυτοί υπεύθυνοι για τις περισσότερες ε, τέτοιες ε, διαδικασίες. Οι δικαστικοί κλητήρες αυτοί δεν ε, είναι καν υφιστάμενοι των δικαστηρίων. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα εναντίον του στο δικαστήριο. Λοιπόν, είχαμε πολλές ε, συναντήσεις ε, στη Βουλγαρία, στο Υπουργικό Συμβουλίο, στη Βουλή. Έχουμε ενημερώσει τους πάντες. Υπάρχει επίσης η υπηρεσία καταπολέμησης της διαφθοράς, ε, την οποία επίσης έχουμε ενημερώσει. Μπορώ να σας δώσω και τα σχετικά έγγραφα για να γνωρίζετε το τι συμβαίνει. Υπάρχει επίσης μια διαδικασία κατά ενός ατόμου στη Βουλγαρία ενός ατόμου ο οποίος ε, ακριβώς ε, είδε την περιουσία σου να ε, πληστηριάζεται ε, όπως επίσης και η δική μου οικογένεια που έμεινε άστεγη. Λοιπόν, θα δώσω τώρα τον λόγο συνάδελφο από, τον, από τη Βάρνα. Κυρίες ε, και κύριοι, σύντομα, το, πρόγραμμα είναι, το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο στην Βουλγαρία. Τα τελευταία χρόνια έχουν αυξήσει τα επιτόκια στα στεγαστικά δάνεια, οι τράπεζες ε, το 2016 μαζέψαμε υπογραφές, ε, όπως επίσης και το 2017 και θέλουμε έτσι να οργανωθεί ένα δημοψήφισμα για να αλλάξει ο αστικός ε, κώδικας. Τα βουλγαρικά ΜΜΕ δεν λένε κουβέντα για την υπόθεση. Εγώ ως δικηγόρος καθημερινά ασχολούμαι με τέτοιες ε, υποθέσεις Δηλαδή καθημερινά οι τράπεζες ε, κινούν τέτοιες διαδικασίες κατά βούλγαρων υπηκών, ε, τις οποίες κερδίζουν. Και δεν φταίνε πάντα οι ενδιαφερόμενοι. Ε, μιλάμε για τις μεγάλες τράπεζες, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, Raiffeisen Bank, Unicredit. Το πρόβλημα είναι πραγματικά μεγάλο, γι' αυτό σας παρακαλώ να κρατήσετε ανοιχτή την αναφορά για να συνεχίσουμε τον αγώνα μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλέσαμε και την μόνιμη αντιπροσωπεία της Βουλγαρίας εδώ, αλλά δεν ήρθανε. Το λόγο τώρα έχει εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν έχουμε αναφερθεί όμως την τελευταία αναφορά ναι, θέλετε και εσείς να πάρετε το λόγο, παρακαλώ. Η κυρία Σβέτλα Μιλάνοβα έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ εκπροσωπώ την Βιολέτα Κοσποντίνοβα, την αναφέρουσα δηλαδή, η οποία δεν παρευρίσκεται εδώ σήμερα. Για μία ακόμα φορά, και ένα φορά αυτή, έχει να κάνει με ζητήματα τα οποία φαίνεται να είναι εντελώς μεμονωμένα, αλλά στην πράξη βλέπουμε ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Η κυρία Κοσπο... Κοσποντίνοβα αναφέρεται εδώ πέρα σε περιστατικά τα οποία πλέον έχουν γίνει συστηματικά στην Βουλγαρία. Βλέπετε πάρα πολλά στοιχεία στο ίδιο το έγγραφο της αναφοράς. Βλέπετε τα προβλήματα τα οποία αντιμετώπισε με τον υπόθηκο δάνειό τη, περίμενε ότι θα είχε ένα επιτόκιο της τάξης του 3%, κατέληξε τελικά να καταβάλει τόκου της τάξης του 12%. Ουσιαστικά είχε αποπληρώσει το ίμιση του δανείου της, και ακολουθήθηκε για το υπόλοιπο ημισή μια εντελώς παράνομη τελικά παράτυπη διαδικασία. Και ουσιαστικά αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι η κοινοτική νομοθεσία δεν εφαρμόζεται πολύ απλά στη Βουλγαρία. Μόνο σε αυτό το συμπέρασμα μπορεί να καταλήξει κανείς. Η τράπεζα, ο πιστωτή, εν προκειμένου, επέβαλε τους όρους του, ενώ ο φιλέτης η κυρία Κοσμποντίνοβα δεν μπόρεσε ουσιαστικά να, καθόλου, τοποθετηθεί καθόλου και βλέπουμε ότι στα πλαίσια του ανυπόθηκου αυτού δανείου υπήρχαν πολλές καταχρηστικές ρήτρε. Και δυστυχώ η κυρία Κοσποντίνοβα δεν γνώριζε για την ύπαρξη των καταχρηστικών αυτών ρητρών, αφού είχε υπογράψει βέβαια τη σύμβαση αυτή. Ουδέποτε ενημερώθηκε, ουδέποτε έλαβε την κατάλληλη πληροφόρηση από την τράπεζα. Η αναφέρουσα λοιπόν δεν είχε την απαραίτητη ενημέρωση, όπως κανονικά προβλέπεται από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Δεν γνώριζε λοιπόν ποια διαδικασία επρόκειτο να ακολουθεί σε περίπτωση μη αποπληρωμής του δανείου. Η αναφέρουσα λοιπόν βρέθηκε σε μια πολύ δινή θέση, δεν χαίρει καθόλου ένδικων μέσων αυτή τη στιγμή προκειμένου να προασπίσει τον εαυτό της. Έχει βρεθεί σε πολύ δινή οικονομική θέση, δεν έχει πλέον πουθενά που να μείνει και βέβαια έχει και εξαρτώμενο παιδί. Και βέβαια έχασε εντελώ και το τμήμα εκείνο του δανείου το οποίο είχε αποπληρώσει. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ε, η διαδικασία εκτέλεσης απαιτήσεων πληρωμή που εφαρμόζει η Βουλγαρία ουσιαστικά δεν συνάδει καθόλου με την ενωσιακή νομοθεσία, αλλά ούτε και η δικαστική απόφαση που ελήφθη από βουλγαρικό δικαστήριο συνάδει με τα όσο προβλέπει ο ευρωπαϊκός νόμος. Τρεις συγκεκριμένα ήταν ε, οι εντολέ συνεργαστικής εκτέλεσης που δημοσίευσε η Βουλγαρική Τράπεζα και πουλήθηκε τελικά μέσω δημοπρασία στο διαμέρισμά τη σε πολύ χαμηλότερη τιμή από την πραγματική του αξία. Καταλαβαίνετε λοιπόν σε τι κατάσταση αναφερόμαστε εδώ πέρα. Ουσιαστικά αναφερόμαστε σε πρακτικές οι οποίες στην πράξη αποτελούν κλοπή. Κλοπή της περιουσίας των ίδιων των ιδιωτών. Πρόεδρο. καταλαβαίνω ότι διανύεται μια πολύ δύσκολη κατάσταση σε προσωπικό επίπεδο, αλλά βλέπουμε ότι το φαινόμενο αυτόν οριζόντιο τουλάχιστον στην Βουλγαρία αφορά και άλλου ανθρώπους. Απευθύνομαι στον κύριο Ματιάκα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχετε το λόγο, μπορείτε να μας παρουσιάσετε την τοποθέτηση Ευρωπαϊκή Επιτροπή επί του ζητήματο αυτού. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και τους αναφέροντες. Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουμε λάβει γνώση του προβλήματος αυτού και μάλιστα και εμεί οι ίδιοι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουμε λάβει απευθεία πολλέ καταγγελίε από ιδιώτες ή από οργανώσει εκπροσώπηση τη κοινωνία των πολιτών στη Βουλγαρία. Καταγγελίε οι οποίε ε, καταδεικνύουν ότι ενδεχομένω να υπάρχει όντω σύγκρουση ε, συμφερόντων ε, ανάμεσα στα όσα ισχύουν στη Βουλγαρία όσον αφορά δηλαδή τις εντολές αναγκαστικής εκτέλεσης και των συμφερόντων των πολιτών. Ενδεχομένως όντως οι πρακτικές αυτές να μην συνάδουν με την οδηγία όσον αφορά τις κατακριστικές ρήτρες των συμβάσεων. Να φέρουμε εδώ πέρα στην οδηγία 93 13 και ενδεχομένω να μην συνάδουν επίση και με την ίδια την ομολογία του Δικαστηρίου τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Οδηγία 93-13 δεν περιέχει διατάξεις όσον αφορά την δικονομία που θα πρέπει να ισχύει σε περίπτωση εντολών αναγκαστικής εκτέλεσης. Πάντως υπάρχει νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει να κάνει με την αποτελεσματικότητα των θεμητών και δίκαιων ρητρών. Μολονότι λοιπόν δεν υπάρχουν διατάξει στο πλαίσιο τη οδηγία, υπάρχουν αρχέ οι οποίε προκύπτουν από την ομολογία του δικαστηρίου, όπω η αρχή τη αποτελεσματικότητα, σύμφωνα με την οποία δεν θα πρέπει οι αποφάσεις των εθνικών δικαστηρίων να φέρνουν σε ιδιαίτερα δεινή σχέση, θέση με συγχωρείτε, τους ιδιώτες, ιδίως όσον αφορά τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων. Μετά από όλες αυτές τις καταγγελίες ξεκινήσαμε το λεγόμενο διαρθρωμένο διάλογο με τις αρχές της Βουλγαρίας. Υποβάλαμε λεπτομερείς ερωτήσεις όσον αφορά τους κανόνες που ισχύουν στη Βουλγαρία, προκειμένου να καταφέρουμε να καταλάβουμε καλύτερα περί τίνος πρόκειται και θέλαμε επίσης να δούμε ποιες είναι οι δυνατότητες που έχουν ε, οι βούλγαροι καταναλωτές προκειμένου να προσφύγουν κατά των εντολών αυτών αναγκαστικής εκτέλεσης. Οι βουλγαρικές λοιπόν αρχές μας απέστειλαν μια λεπτομερή απάντηση. Ωστόσο, δεν πρότειναν καμία απολύτως αλλαγή και τροποποίηση στους υφιστάμενους κανόνες. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο οι υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής πολύ πρόσφατα απέρριψαν την απάντηση αυτή των βουλγαρικών αρχών και επομένως τώρα θα πρέπει να δούμε ποια είναι τα επόμενα βήματα τα οποία θα μπορούσαμε να κάνουμε στο ζήτημα αυτό. Έτσι έχει πάνω κάτω η κατάσταση και αυτή είναι η ανάλυση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τουλάχιστον. Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε πολύ. Τώρα το λόγο έχουν οι συνάδελφοι για τυχόν παρεμβάσεις. Ο κύριος Μάλινοφ έχει το λόγο. Πολύ φοβάμαι ότι θα αναρωτιέστε πώς τα βουλγαρικά δικαστήρια μπορεί να είναι τόσο αδύναμα. Ενδεχομένω θα αναρωτιέστε για ποιο λόγο μετά από τόσα πολλά χρόνια κατάχρηση εξουσία από τι τράπεζε Τίποτα δεν έχει συμβεί στην πράξη. Μία απάντηση μόνο μπορώ να δώσω. Και θα πρέπει να είμαι απόλυτα ειλικρινή μαζί σα. Τα βουλγαρικά δικαστήρια είναι πραγματικά αδύναμα. Πολύ φοβόμαστε ότι ε, ουσιαστικά μπορεί να επηρεαστούν από πολιτική επιρροή, από την επιρροή των επιχειρήσεων και γι' αυτό το λόγο βρισκόμαστε υποκαθεστώς παρακολούθησης μαζί με τη Ρουμανία. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι όταν προσχωρήσαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπήρχε ένας κλάδος, ο δικαστικό, ο οποίο είχε θεωρηθεί τότε ότι δεν είχε περάσει από αρκετέ μεταρρυθμίσει και μεταρρυθμίσει αυτέ ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί και υπάρχουν πολλοί πολίτε, είτε στη Βουλγαρία είτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που αυτή τη στιγμή έχουν να αντιμετωπίσουν μια αναποτελεσματική δικαστική αρχή ή πολλέ φορέ αναποτελεσματικέ δικαστικέ διαδικασίε. Και αυτό αποτελεί πραγματική τραγωδία. Πάρα πολλοί είναι οι πολιτικοί, όλοι οι πολιτικοί βασικά στη Βουλγαρία γνωρίζουν πώ έχει το, το θέμα. Πολλοί είναι οι πολίτε που γνωρίζουν πώ έχει κατάσταση και έχουν γίνει και πάρα πολλέ διαδηλώσει. και πολλοί έχουν βρεθεί στην κατάσταση που περιέγραψαν ε, οι αναφέροντε. Α δούμε λίγο τη νομική βάση, τη νομική πτυχή. Βλέπουμε ότι ακόμα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και δεν είμαι καθόλου σαρκαστικό τώρα, αλλά πρέπει να το πω αυτό, ακόμα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακόμα διερευνά το βουλγαρικό δικαστικό σύστημα. Και μα λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και την παραθέτω τώρα, επιβεβαιώνει ότι οι δικονομικές αρχές της Βουλγαρίας ενδεχομένως όντως να επιτρέπουν σε κάποιους πιστωτές της Βουλγαρίας να προωθούν διαδικασίες fast track όσον αφορά τις εντολές συναγκαστικής εκτέλεση. Ότι καταφέρνουν δηλαδή και επισπεύουν αυτέ τι διαδικασίε. Δεν είναι, το σύστημα, το σύστημα δυσχεραίνει την κατάσταση των Βουλγάρων υπηκών, ότι ουσιαστικά διευκολύνει την κατάσταση όσον αφορά τις αρμοδιότητες που έχουν οι ίδιες οι τράπεζες. Νομίζω λοιπόν ότι δεν μπορούμε να προσπιστούμε σε καμία περίπτωση δημοσίως αυτές τις πρακτικές. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο ζητώ αναφορές αυτές να παραμείνουν ε, ανοιχτές, αλλά παράλληλα νομίζω ότι και η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών θα πρέπει να γνωμοδοτήσει για αυτές τις αναφορές. Μα ουσιαστικά πρόκειται για πραγματικέ τώρα υποθέσει που δεν υπάρχει πραγματική νομική υπεράσπιση των πολιτών σε εθνικό επίπεδο και δεν είναι τυχαίο ότι έχουμε αναφέροντε από τη Βουλγαρία εδώ σήμερα. Δεν θα έλεγα ότι ακούγονται απεγνωσμένοι, πάντως σε κάθε περίπτωση σας εγγυώμαι ότι έχουν εξαντλήσει κάθε δυνατότητα στη Βουλγαρία και σίγουρα οι δικηγόροι του κάναν κάτι το δυνατό. Αφού εξαντλήσαν λοιπόν όλε τι δυνατότητε που είχαν σε εθνικό επίπεδο, ήρθαν εδώ πέρα. Θεωρώ λοιπόν θα πρέπει να ζητήσουμε γνωμοδότηση από την Επιτροπή Εσωτερική Αγορά και να επενθυμίσουμε στου πολίτε τη Βουλγαρία ότι οποιοδήποτε και αν είναι το νομικό σύστημα τη χώρα του, υπάρχουν και άλλε δίωδοι μέσω τη Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ενδεχομένω από νομική πλευρά να μην είμαστε πάρα πολύ ισχυροί, αλλά είμαστε πάρα πολύ ισχυροί όσον αφορά τη δημόσια προβολή των υποθέσεων αυτών και την επιρροή τη κοινή γνώμη. Σα ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Κούνεβα, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, αυτό τον τρόπο που θα δώσουμε σήμερα εμεί σαν απάντηση στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι Βούλγαροι πολίτε θα εξαρτηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό η πιστοσύνη στην Ευρώπη και στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Γιατί <clears throat> είναι εκατοντάδες, χιλιάδες οι Βουλγαροί πολίτες που έχασαν την περιουσία τους χωρίς καν να το καταλάβουν με διαδικασίες κατάσχεσης εξπρές ή άλλοι που αντιλήφθηκαν ξαφνικά ότι τα επιτόκια των δανείων τους είχαν αυξηθεί χωρίς να το καταλάβουν. Επιπλέον, Έχουμε και ένα άλλο πρόβλημα το οποίο είναι επίσης τόσο βαρύ. Ότι όταν πια έχουν κάνει την κατάσχεση των πυρουσίων και πολλάνε σε κάποιο άλλο πολίτη την πυρουσία αυτή και δεν, δεν παίρνουν τα χρήματα τα οποία α, χρωστάει στο δάνειο ο πολίτης αφού πούλησαν τα ακινητά όλα, απαιτούν από το πολίτη και άλλα χρήματα επιπλέον. Α πούμε ήταν 8 εκατομμύρια, το πούλησε 6. Ακόμα 2 εκατομμύρια ζητάνε από το πολίτη. Αφού πούλησαν όλα. Α, απαιτούν ακίνητα των γονιών τους, των παππούδων και ελιάδων. Αυτό είναι παράδεκτο και παράνομο. Η, η απάντηση της Επιτροπής δεν είναι ουσιαστική και προτείνω, η αφορά, οι αφορές όλες να μένουν ανοιχτές, προτείνω να οργανωτούμε και να πάμε στη Βουλγαρία, να μιλήσουμε και με τα κινήματα, γιατί μαζεύουν πάρα πολλές πολίτες υπογραφές, με πολλοί οργανισμοί και δικαστήρια να συζητήσουμε μαζί τους και με την κυβέρνηση, να καλέσουμε όμως εκπρόσωπους της Επιτροπής της Ευρώπης και να καλέσουμε και από την ΙΜΚΟ συνάδελφοι οι οποίοι να συμμετέχουν και να δούνε πώς διαχειρίζεται η εσωτερική αγορά στη Βουλγαρία, πόσο πολύ παρανομούν και πόσο σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι Βουλγαροί πολίτες. Σας ευχαριστούμε πολύ. Απευθύνομαι για άλλη μια φορά τώρα στους αναφέροντες. Έχει το καθένας από ένα ή δύο λεπτά για να δευτερολογήσετε. Έχετε το λόγο. Starting out in the same order as Ακολουθήσουμε την ίδια σειρά όπως και πριν. Φιλίποβα πρώτη, κυρία Φιλίποβα. Искам да кажа, че проблема с потребителската защита в България допълнително. Ευχαριστώ πολύ. Το πρόβλημα αυτό επίσης επιβαρύνεται γιατί δεν υπάρχει νόμος για την χρεοκοπία φυσικών προσώπων. Είμαστε η μόνη χώρα στην οποία εξακολουθούν τα χρέη να παραμένουν επάπειρον και θα ήθελα να πω το εξής. Έχω εντωμεταξύ διαπιστώσει πως η Societe General στην Βουλγαρία έχει πολύ, υψηλότερους, πολύ ψηλότερα επιτόκια για τους βούλγαρους πελάτες από ότι τα επιτόκια στη Γαλλία και όπως είπαμε υπάρχει μια διαφορά ε, μεταξύ των επιτοκίων στην αρχή του δανείου και μετά τα επιτόκια ανεβαίνουν και βεβαίως αυτό δυσκολεύει την ζωή κυριολεκτικά των πέλατων. Ουσιαστικά οι τράπεζες ε, αφαιρούν την περιουσία ή την αγοράζουν μέσω κάποιων θηγατρικών τους επιχειρήσεων και τα κέρδη πάλι πάνε στα ταμεία των τραπεζών. Δεν υπάρχουν στατιστικά στοιχεία και επίσημα έγγραφα αλλά νομίζω αυτό μπορούμε να το αποδείξουμε σε μια τακτική διαδικασία στο δικαστήριο. Και βεβαίως ε, είμαστε σε επαφή με τους βουλευτές μας, αλλά παρόλα αυτά δεν πετύχαμε τίποτα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσατε τον λόγο. Όλοι εμείς ήρθαμε εδώ με μια μεγάλη ελπίδα δηλαδή να μας στηρίξουν οι ευρωβουλευτές γιατί τα θεσμικά όργανα είναι διεφθαρμένα στην Βουλγαρία μας έχουν απογοητεύσει και έχουμε χάσει κάθε ελπίδα ότι μπορεί να αλλάξει κάτι γι' αυτό σας παρακαλώ εσάς προσωπικά και εξ ονόματος ε, των ε, συντρόφων μου εδώ να δείτε το πρόβλημα μας. Πραγματικά πρέπει να ζητήσετε από την Κομισιόν να υπάρξει ένας μηχανισμός ε, ελέγχου και να ξαναδεί το θέμα των βουλγαρικών δικαστηρίων για να μπορέσει να αλλάξει ο νόμος. για να ολοκληρωθεί επιτυχώς αυτή η υπόθεση χωρίς ε, την δική σας ε, την παρέμβαση δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε τίποτα και κανένας βουλγαρος πολίτης δεν θα μπορέσει να πάρει πίσω την περιουσία του. Κυρίες και κύριοι, ο ευρωπαϊκό λαός εμπιστεύεται το ευρωπαϊκό δίκαιο και τις ευρωπαϊκές αξίες και από όταν προέκυψε αυτό το πρόβλημα είναι πραγματικά φόρητο και το μεταξύ χάνουμε και την εμπιστοσύνη μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί στην Ευρωπαϊκή Ένωση βασιστήκαμε ακριβώς για να υπάρξει μια προστασία των πολιτών. Έχουμε κάνει ό,τι μπορούμε με τα δημοκρατικά μέσα, διαμαρτυρίες, διαδηλώσεις, συζητήσεις με τους βουλευτές πρωτοβουλίες πολιτών. Αλλά τα ΜΜΕ, τα κόμματα δεν μας στήριξαν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και οι κυβερνώντες ε, στην Βουλγαρία προφανώς δεν θέλουν να αλλάξουν τους ε, νόμους. Και παρακαλώ ακριβώς ε, να λάβετε το θέμα αυτό γιατί εντωμεταξύ η ατμόσφαιρα είναι επαναστατική. Ο κόσμος χάνει τα σπίτια του. Μία μικρή συμπλήρωση από εμένα. Εμεί οι Βούλγαροι είμαστε Ευρωπαίοι πολίτες και θέλουμε να ισχύσει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για να προστατεύονται και οι Βούλγαροι καταναλωτές όπως οι Ευρωπαίοι. Να σας πω, εγώ είμαι επικεφαλής ε, του κινήματος βουλγαρών πολιτών. Θέλω να σας παρακαλώ να μην ανοιχτή η αναφορά, γιατί ε, ήδη 70 ειδικοί εργάζονται ε, σε συνεργασία με το Βουλγαρικό Κοινοβούλιο. Γι' αυτό σας παρακαλώ να αφήσετε ανοιχτή την αναφορά έτσι ε, ώστε να αλλάξει το νομικό πλαίσιο στην Βουλγαρία. Αυτή τη στιγμή η βουλγαρική νομοθεσία δεν ανταποκρίνεται σε ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Δεν υπάρχει ισότητα μεταξύ των βουλγαρών πολιτών. δεν έχουμε τη δυνατότητα να αποδείξουμε την αθωότητά μας. Σε μένα προσωπικά επιτέθηκαν, επιτέθηκαν στον σύζυγό μου, προσπάθησαν να τον σκοτώσουν. Έτσι έχουν τα πράγματα. Και ακριβώς ε, τώρα προσπαθεί η ολιγαρχία να σοπάσει όσους κάνουν κάτι για τα δικαιώματα των πολιτών. Πρόεδρο, σε ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να συνοψίσω. Όπως γνωρίζουμε λοιπόν από αυτό που ακούσαμε σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί οριστικά να αποφασίσει μια που συνεχίζεται ο διάλογος. Όμως, εμείς περιμένουμε να μας στείλετε μια έκθεση γραπτά, έτσι, πρέπει συνέχεια να αναφέρεστε σε εμά με ό,τι νέο υπάρχει. Αυτό θα το εκτιμήσουμε πολύ. Λοιπόν, τι πρέπει να προσέξουμε. Το θέμα της λογοδοσίας των βουλγαρικού συστήματος και κατά πόσο συνάδει με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία ε, για τους καταναλωτές. Είχαμε στραφεί στην ΕΜΚΟ και νωρίτερα και είχαμε ζητήσει γνωμοδότηση. Εμάς δεν μα την έχουν δώσει ακόμα αυτή τη γνωμοδότηση, αλλά μέσω τη γραμματεία θα του το ξαναζητήσουμε να το κοιτάξουν αυτό το θέμα. Ελπίζουμε να την ετοιμάζουν την απάντησή τους, γιατί είναι και αυτό ένα στοιχείο που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας για να αποφασίσουμε. Λοιπόν, αφού συνεχίζεται ο διαρθρωμένος διάλογος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι έρευνες. Και στο τέλος της διαδικασίας αυτής ελπίζω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κοιτάξει και να μελετήσει σε βάθος τις δικαστικές αποφάσεις και υπό το φως του άρθρου 47 ε, της Χάρτας Θεμελιωμένων Δικαιωμάτων να μας δώσει μια απάντηση. Και σε εσά τους αναφέροντες θέλω να σας μεταφέρω το μήνυμα της Επιτροπής μας. Αυτά τα οποία μας παρουσιάσατε μας απασχολούν και μας ανησυχούν πολύ. Οι Βούλγαροι πολίτες θα έπρεπε να μπορούν να συνεχίσουν να εμπιστεύονται το Ευρωπαϊκό Σύστημα Δικαιοσύνης και την Επιτροπή αυτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και όλες τις αρχές στις οποίες βασιζόμαστε. Αυτό θα κάνουμε και θα συνεχίσουμε. Και πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ταξιδέψατε για να έρθετε ως εδώ. Εποφεληθείτε λίγο από τη διαμονή σας εδώ στις Βρυξέλλες και καλό ταξίδι πίσω στη Βουλγαρία. Σας ευχαριστούμε. Τώρα ε, ρωτάω τους συναδέρφους να μου πούν αν συμφωνούν. Θα μείνει ανοιχτή λοιπόν η αναφορά. Θα περιμένουμε τις πληροφορίες που ελπίζουμε να μας στείλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά θα στείλουμε και επιστολή, εγώ τουλάχιστον αυτό θα ήθελα στις βουλγαρικές αρχές και να ερευνήσουμε και με την ΙΜΚΟ παρετέρω. Μήπως μπορούμε να καταλήξουμε σε κάτι. Είναι πήγον το ζήτημα. Λοιπόν, συμφωνούμε. Καλώς. Ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζουμε. Το σημείο 16 το εξετάσαμε ήδη, οπότε πάμε στο σημείο 17 που είναι η αναφορά 11-19 για εικαζόμενη διάκριση σε βάρος φοιτητών εξαιτίας του Βρετανικού συστήματος. Ο αναφέρον είναι εδώ. Ο ένας, όλος δεν θα έρθει. Δανάη, δεν θα έρθει σήμερα ή έρχεται. Όχι, α, δεν είναι εδώ. Ωραία. Θα δώσω λοιπόν το λόγο σε εσά, κύριε Μάρκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα αρχίσω παρουσιάζοντας κάπως σύντομα, περιγράφοντας τα δικαιώματα των ε, Ευρωπαίων πολιτών βάσει της οδηγίας 3814 ε, και λέει ο, το άρθρο 24 ότι όλοι όσοι κατοικούν ε, στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια έχουν την ίδια μεταχείριση με τους ε, υπήκους της εν λόγω χώρας, χωρίς διακρίσεις και ότι το δικαίωμα αυτό διευρύνεται και σε μέλη της οικογένειας ακόμα και αν δεν είναι Ευρωπαίοι υπήκοοι. Και αυτό έχει ακολουθήσει και το δικαστήριο όσον αφορά την πρόσβαση ε, στην εκπαίδευση, για δίδακτρα κτλ. Ως εξαίρεση στην παράγραφο αυτή, οι χώρες μέλη δεν είναι υποχρεωμένες πριν να υπάρχει μόνιμη διαμονή να προσφέρουν τέτοια επιδόματα επιχορηγήσεις και τα λοιπά σε μέλη της οικογένειας. Άρα δεν μπορούν να παρεκκλίνουν από τον κανόνα της ίσης με εξαίρεση αυτές τις περιπτώσεις. Εργάζεται ε, στην, σε χώρα μέλος ο αναφέρον, οπότε υποφελείται κανονικά από την ίση μεταχείριση όπως όλοι οι εργαζόμενοι και αυτό θα πρέπει να ισχύει και για τον σύντροφό του. Βάσει της λόγω νομοθεσίας του 2011 που εφαρμόζεται στην Αγγλία, οι εργαζόμενοι μπορούν να έχουν τέτοια οικονομική στήριξη μόνο εφόσον κατοικούν στην ε, επικράτεια που έχουμε συμφωνήσει τρία χρόνια πριν. Και είναι ε, κάτοικο στην πρώτη μέρα του ακαδημαϊκού έτους. Προκειμένου να έχει αυτή την οικονομική στήριξη ένας ε, Ευρωπαίος υπήκος πρέπει να υπακούει και στους κανόνες περί διαμονής. Η εκτίμηση Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ότι παρόλο που είναι ευνοϊκή η διάταξη, πρέπει να πούμε ότι ο γεωγραφικός χώρος που λαμβάνεται υπόψη ως ε, κατοικία διαμονής είναι εκείνος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Οπότε, αν βάλουμε επίση όλου του πολίτε, θα πρέπει να ισχύει ότι ισχύει και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αν όμω τελικά η υπάρχει αυτή η απέτηση για τα τρία χρόνια και αυτό ισχύει για όλους ανεξάρτητα της υπηκότητας, ακόμα δηλαδή και σε υπηκόους του Ηνωμένου Βασιλείου, τότε δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει διάκριση. Δικαιολογείται από την ομολογία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα σας ε, υποβάλει γραπτή έκθεση πάνω σε όλα αυτά και εκεί θα παρουσιάζουμε περισσότερες λεπτομέρειες στην θέση μας. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Συζήτηση τώρα. Οι συνάδελφοι, παρακαλώ. Η Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ πολύ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Από ό,τι καταλαβαίνω, ο αναφέρον ζητάει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την άποψή της όσον αφορά τη Βρετανική νομοθεσία. Και αυτό έκανε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οπότε νομίζω ότι μπορεί να κλείσει αναφορά. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να αναλάβουμε οποιαδήποτε άλλη δράση εφόσον δεν υπάρχει διάκριση. Ευχαριστώ. Πολύ καλή πρόταση κατά τη γνώμη μου. Και εγώ πιστεύω ότι αυτό πρέπει να κάνουμε είναι να περιμένουμε τη γραπτή απάντηση και νομίζω ότι πρέπει να το στείλουμε και στην ομάδα steering για το Brexit, να το δούνε και εκείνοι, να ξέρουν ποιες είναι οι διατάξεις που ισχύουν και ποια είναι η κατάσταση δεδομένου του επερχόμενου Brexit. Και μετά να την κλείσουμε, να περιμένουμε την απάντηση της Επιτροπής και να κλείσει, να πάει και στο Brexit σας είπα. Πίτερ. Σωστά τα είπατε κυρία Πρόεδρε. Εδώ στα χαρτιά μου βλέπω ότι αναφορά έχει σταλεί και στην Επιτροπή Πολιτισμού και πρέπει να υπενθυμίσουμε ε, ότι ε, εδώ πέρα δηλαδή μου γράφουν ότι πρέπει να σταλεί προς ενημέρωση και στην Επιτροπή Προϋπολογισμού ε, οπότε να το κλείσουμε το, το πακέτο με τις απαντήσεις όχι όχι Πίτερ τα στείλαμε μόνο προς ενημέρωση δεν τους ζητήσαμε να κάνουν κάτι Είπαμε να ενημερώσουμε και την ομάδα steering για το Brexit, τίποτα άλλο, για ενημέρωση και μετά θα το κλείσουμε λοιπόν. Ωραία, με το χρόνο καλά τα πάμε. Μπορούμε να σταματήσουμε τώρα, τελειώσαμε. Για σήμερα το πρωί. Θα τα ξαναπούμε στις 2.30. Οπότε έχετε μεγάλο διάλειμμα για να φάτε και φροντίστε μια που έχετε περισσότερο χρόνο να χαμογελάσετε και λίγο περισσότερο.